εξαχθεί αύριο. Περνάμε στο επόμενο θέμα, το τελευταίο για σήμερα, την έκθεση Πέτρη Γέζεκ με θέμα το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση. Το λόγο έχει πρώτα για τέσσερα λεπτά ο εισηγητής ο κύριος Πέτρη Γέζεκ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι. 1,5 χρόνο μετά τη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Κεφαλαιαγορές, έχουμε επιτέλους ένα αυτό παράδειγμα για το πώς θα το διαμορφώσουμε. Προτείνεται εξυγχρόνιση της οδηγίας, εξυγχρονισμός της οδηγίας για το ενημερωτικό δελτίο, ώστε να μπορέσουν να ενημερώνονται καλύτεροι επιχειρήσεις, Ένονται τα, οι ρυθμιστικές για τι μικρές ε, εταιρείε ή για τα μικρά ποσά και στηρίζονται ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτού του στόχου και προτείνει πολλές καινοτομίε, ώστε να γίνει ε, η σχετική νομοθεσία πολύ πιο κατάλληλη και να ανταποκρίνεται στις, στις ανάγκες. Για παράδειγμα, αυξάνονται κατώτατα όρια για τις εξαιρέσεις από, το, από τις ρυθμίσεις. Επίσης, έχουμε μια εξαίρεση για το Ευρωπαϊκό Ενημερωτικό δελτίο και διευκόλυνση των ε, επιχειρήσεων για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Χάρη στις διαπραγματεύσεις επί Σλοβακικής Προεδρίας ε, τελειοποίησαμε τις ε, θέσεις μας και καταλήξαμε σε συμφωνία που ευελπιστώ ότι θα εξυπηρετήσει όλους τους εκδότες που θέλουν να βρουν κονδύλια στις αγορές. Για παράδειγμα, αυξήσαμε ε, σε ένα εκατομμύριο το ποσό για να παρέχεται εξαίρεση από τα κριτήρια του κανονισμού. Έτσι θα, θα γίνεται πιο εύκολη χρηματοδότηση και θα μπορούν οι επιχειρήσεις ε, να δανείζονται χωρίς υπερβολικές γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Επίσης, ε, με το ενημερωτικό δελτίο για την ανάπτυξη ε, μειώνεται το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν διασυνοριακά να δανειστούν και επίσης ε, το Ευρωπαϊκό Ενημερωτικό Δελτίο για την Ανάπτυξη θα βελτιώσει την πρόσβαση στο κεφάλαιο μικρότερων εκδοτών προκειμένου να αναζητήσουν χρηματοδότηση από τις κεφαλαίες αγορές. Αυτό να, υπερβα... να στηρίζονται υπερβολικά και να από, τις... από την τραπεζική χρηματοδότηση. Επίσης, με το νέο καθεστώς θα μειώσουμε το κόστος για τους εκδότες και θα αυξήσουμε την ε, σημασία και το ευανάγνωστο των πληροφοριών ε, για τους επενδυτές. Έτσι θα έχουμε αύξηση και ενίσχυση και της ε, προστασία των επενδυτών. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουν δευτερογενεί εκδόσει οι ε, επιχειρήσει με εξορθολογισμένη διαδικασία. Ελαχιστοποιούμε τι εθνικέ εξαιρέσει και τη διακριτική ευχέρεια, αυξάνοντα την εναρμόνιση και ενισχύοντα τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Κατά τη γνώμη μου, ε, αυτό το νόημα θα πρέπει να έχει Ένωση Κεφαλαιογορών. Χρειαζόμαστε εναρμονισμένα μέτρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, να μειώσουμε τι γραφειοκρατικέ διατυπώσει για τι ε, μικρέ επιχειρήσει, να εξασφαλίσουμε προστασία του επενδυτή και επίση ε, να ενισχύσουμε τη χρηματογορά στην Ευρώπη, να διευκολύνουμε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση με πρόσβασή του στι κεφαλαιογορέ. Κάτι τέτοιο θα ενισχύσει ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία και θα ε, μα αυξήσει την ανάπτυξη, κάτι που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα σε αυτού του αβέβαιου και χαλεπούς καιρού. Ευχαριστώ κατακλείδη του και ηγητές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Σλοβακική Προεδρία για την εργόδη προσπάθειά του και την αφοσίωσή του υπέρ της ολοκλήρωσης αυτής της φιλόδοξη μεταρρύθμισης ε, του ρυθμιστικού πλαισίου για το ενημερωτικό δελτίο. Σα ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Τώρα εκ μέρου Ευρωπαϊκής το λόγο έχει ο αντιπρόεδρο Βάλντι Ντομπρόφσκης. Αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Βεβαίως η οθέτηση της πολιτικής συμφωνίας θα είναι σημαντικό βήμα επιτρέποντας διασυνορικές επενδύσεις, ε, δίνοντας τις επιχειρήσεις ευκολότερο τρόπο να αντλήσουν από τις κεφαλαιγορές και να έχουμε πληροφορίες για τους επενδυτές. Η αναθεώρηση των κανόνων για το ενομηρωτικό δελτίο είναι κάτι σημαντικό. Μετά από 12 χρόνια εναρμονισμένων κανόνων, θα πρέπει ε, να αναθεωρηθεί ε, το, η διαδικασία. Ε, ακούσαμε τους εκδότες, επενδυτές, τους διαχειριστές της αγοράς μετά την τελευταία μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα το 2010. Οι νέοι κανόνες θα εισαγάγουν ένα νέο ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορεί να βασιστούν οι επενδυτές σε ένα νέο ε, ε, μια νέα διαδικασία εγγραφής επίσης για δευτερεύουσες εκδόσεις. Θα ήθελα να παρουσιάσω τα βασικά θετικά σημεία ε, του ε, νέου ε, κανονισμού. Το ενημερωτικό δελτίο θα επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλούν κεφάλαιο, χρησιμοποιούν λοιπόν το ενημερωτικό δελτίο για το σκοπό αυτό. Πάρα πολλές αγορές σήμερα μπορούν να γίνουν ε, ε, αγορές ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το μέλλον. Ε, το νέο όριο θα, θα είναι 8 εκατομμύρια σε σχέση με το όριο το προηγούμενο. Μπορούν τα κράτη-μέλη να βασιστούν στις κανόνες τους εθνικούς προσφοράς για να ε, αναπτύξουν τις δυνατότητες για μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Θα ωφεληθούν νομίζω όλοι από ένα απλουστευμένο ενομερωτικό δελτίο για τις δευτερεύουσες εκδόσεις. Ε, θα πρέπει οι επιχειρήσεις αυτές να είναι γνωστές στην αγορά όλες τα ενομερωτικά δελτία για τις, με τους μετοχικούς τίτλους θα περιλαμβάνονται εκτιμούμε την εξοικονόμηση για τους εκδότες για 130 εκατομμύρια κατέτος. Τέλος, η εισαγωγή ενός, μιας εγγραφής, ενός ενιαίου ε, εγγράφου. Έχουμε τις ε, πέντε ημέρες αντί για δέκα ημέρες και αυτό θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο και θα επιτρέψει ε, πρόσβαση ε, σε μικρότερο χρόνο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την εξαιρετική εργασία που έγινε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ ε, τον κύριο πίτροπο. Τώρα λοιπόν εκ μέρους του ΕΛΚ ο κύριος Τόμ Βαντεν Καντελάρε. Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει την μεγαλύτερη της αγορά. και μπορούμε τώρα είτε να φοβηθούμε είτε αυτό να το εκμεταλλευτούμε ως ευκαιρία για να προχωρήσουμε περισσότερο στη δημιουργία της ε, κοινή ε, ενωσιακής κεφαλαγοράς. Χρειαζόμαστε επενδύσει αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα. Αυτή λοιπόν η οδηγία είναι σημαντική γιατί σήμερα επιχειρήσει εξαρτώνται από την τραπεζική χρηματοδότηση. Μόνο το 20% των επιχειρήσεων ε, αντλεί χρήματα από την κεφαλαγορά. Έτσι λοιπόν δεν τη χάνει πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων ανάπτυξης που βρίσκεται στις κεφαλαγορές. Σήμερα για τις μικρές επιχειρήσεις το να κάνουν ένα βήμα στην κεφαλαγορά, αυτό το βήμα είναι πολύ μεγάλο. Επίσης τα δελτία, τα ενημερωτικά έχουν γίνει μεταξύ τηλεφωνική κατάλογη και οι επενδυτέ που ενδιαφέρονται δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Οι νέες λοιπόν διατάξεις καθιστούν τα ενημερωτικά δελτία ε, πιο απλά, πιο φτηνά και υπάρχουν ε, και δυνατότητες ε, για επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, για μικρούς εκδότες μέχρι 20 εκατομμύρια. Υπάρχει λοιπόν ένα ε, πολύ πιο εύχριστο ενημερωτικό δελτίο. Έχουμε πολλές εταιρείε οι οποίες θέλουν να απευθυνθούν στην αγορά για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και θα καταφύγουν σε αυτές τις διατάξεις. Κυρίε και κύριοι, αυτός ο νέος κανονισμός προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν αυτές να αντλήσουν κεφάλαια από την αγορά. Αλλά ε, όμως ε, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε εκεί. Πρέπει να υπάρξουν και αλλαγέ όσον αφορά τι πτωχεύσει, τι χρεοκοπίε. Ε, στην Επιτροπή ΕΚΟΝ πρέπει να τα θίξουμε αυτά. Όπω επίση και το να υπάρχει μια ουσιαστική, πραγματική κεφαλαγορά στην Ευρώπη. Η συζήτηση για μια πανευρωπαϊκή αρχή ρυθμίση πρέπει κάποτε να γίνει. Αύριο θα ε, άρουμε το πρώτο εμπόδιο και γι' αυτό πρέπει να υπεψηφίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς ε, πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζήλ ε, και Αγαπητέ Πρόεδρε, καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Γέζεκ, για την έκθεσή του, γιατί ξέρετε για μένα και για την ομάδα μου αυτή η έκθεση καλύπτει πολλές από τις προτεραιότητές μας. Μειώνεται το νομικό κόστος, γραφειοκρατία, ο κατακαιρματισμός, κλειδωμένη ρευστότητα για θεσμικούς επενδυτές, εναρμόνιση των κανόνων Μία λοιπόν βασική πρόταση που η δική μου η ομάδα ήθελε οπωσδήποτε να ε, περάσει ήταν αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν ένα ενιαίο τυποποιημένο έγγραφο για να αντλήσουν κεφάλαια. Και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Με ένα απλό έγγραφο μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να ακολουθήσουν μια εύκολη διαδικασία για να αντλούν κύματα από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το νομοθέτημα θα επιτρέψει το crowdfunding ε, συνεργατικό, στη συνεργατική χρηματοδότηση, η δυνατότητα δυνατότητες που υπάρχουν, υπάρχουν πολλές στην κεφαλαία αγορά, αλλά είναι επίσης σημαντικό ε, όσοι καταφεύγουν ε, και οι τρίτες χώρες μάλλον να μπορούν και αυτές να έρθουν στις ευρωπαϊκές αγορές. Τα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα, μπορούν, θα πρέπει να μπορούν να επενδύουν. Επειδή έχουμε την αποχώρηση του Ρωμαίου Βασιλείου, θα ήταν επιζήμιο ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην υπάρχουν ευέλικτες αγορές. Αυτές βασίζονται κατά 60% στις ευρωπαϊκές κεφαλαγορές. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις θέσεις απασχόλησης, για την ανάπτυξη της Ευρώπης των 27. Ως εκ τούτου, η βελτίωση των δελτίων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γιουτζίλ εκ μέρους ε, της GUNGL. Το λόγο έχει ο κύριος Μιγγέλ Βιέγας. Η πρόταση οδηγίε για το ενημερωτικό δίκτυο αποτελεί ένα βήμα προκειμένου να ε, υλοποιηθεί η Ένωση Κεφαλαγορών. Ε, θέλουμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ε, πρόσβαση κεφαλαγορές μέσω δημόσιων προσφορών κινητών αξιών ή εισηγμένων ε, ή εισαγωγών κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές. Δυστυχώς η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα των χωρών μας. Ε, γιατί η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσει, πιστεύετε θα έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους χρηματοδότηση παρά τις ε, αφιβολίες που υπάρχουν για τις ε, δευτερεύουσες ε, εκδόσεις ή για τις διατυπώσεις που ισχύουν δεν νομίζω ότι συνάδουν με τις προτεραιότητε τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό που χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι ένωση κεφάλαιο αγορών, αλλά πρόσβαση σε δανεισμό και κυρίως δημόσια κονδύλια και προγράμματα για την πρόθεση τη απασχόλησης και τη καινοτομία. και μια πολιτική αναβάθμιση των μισθών που θα βελτιώνει την καθημερινότητα των νοικοκυριών και θα αποκαθιστούν την οικονομία τους στι επιχειρήσει και στην την εμπιστοσύνη του στι επιχειρήσει και την οικονομία. Σας ευχαριστούμε κύριε Βιέγκας. Εκ μέρους των Πρασίνων τώρα το λόγο ο κύριος Ουρτασούν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή, τον κύριο Γιάζεκ, για την πολύ αγαστή συνεργασία που είχαμε. Αύριο οι πράσινοι δεν θα, υπερψηφίσουν αυτή την αναθεώρηση της οδηγίας. Θα κρατήσουμε στάση αποχής, γιατί θεωρούμε το, το πλαίσιο που προτείνει για την απλούστευση είναι υπερβολικά περίπλοκο και έτσι μειώνουμε την προστασία των καταναλωτών ε, για το με την εφαρμογή του ενημερωτικού δελτίου. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, ε, εισηγητή και να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί στα σημεία 7 και 16 προβλέπεται υποχρέωση όλων των εκδοτών να επισημαίνουν υπό συνθήκες ε, μπορούν να εφαρμόσουν bail-in σε ορισμένα τέτοια προϊόντα με βάση την ε, οδηγία για την ανάκαμψη και εξηγέση των τραπεζών. Γι' αυτό ακριβώ δεν θα καταψηφίσουμε, επειδή συμφωνούμε με αυτά τα δύο σημεία. Είναι πολύ θετικέ αυτέ οι δύο παράγραφοι 7 και 16 και αυτό θα μα οδηγήσει να μην καταψηφίσουμε, απλώ να κρατήσουμε στάση αποχή στην αυριανή ψηφοφορία. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία για τον κανονισμό ε, για το ενηματρικό δελτίο είναι πρόοδος και θα ήθελα να συγχαρώ ε, τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές και τις συζητήσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά τη διάρκεια των τελευταίων μήνων για να είναι πιο απλό για τις επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρομισές επιχειρήσεις να αντλούν κεφάλαια από τις αγορές και να εισάγονται στο χρηματιστήριο μπορεί να εξασφαλίσει ευημερία και ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις έχουμε, βασιζόμαστε πολύ στην άντληση κεφαλαίων από τις ε, τράπεζες. 25% μόνο προέρχεται από τις ε, αγορές κεφαλαίων. Στις Ηνωμένε Πολιτείε είναι το αντίθετο, γι' αυτό θα πρέπει να εμβαθύνουμε ε, στις κεφαλαιοχωρές με το καθεστώς αυτό του ενομερωτικού δελτίου θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αντλούν κεφάλαια με βάση ένα κοινό πλαίσιο υπάρχουν Βεβαίως από την προηγούμενη οδηγία πράγματα που έχουν απομείνει. Ε, η προηγούμενη οδηγία δεν επέτρεψε μια καλή ε, λειτουργία ενιαίας αγοράς και δημιουργούσε κάποια βεβαιότητα νομική και μερικές επιβαρύνσεις που ε, αύξαναν το κόστος και ήταν, υπήρχαν και ανεπάρκειες. Πολλοί μετέφεραν την οδηγία εθνικά σε 28 διαφορετικά καθεστώτα. Καλύτερα να έχουμε έναν κανονισμό με εναρμονισμένους κανόνες και αυτό είναι αναγκαίο. Βεβαίως χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα συστήματα για τους συνήθεις χρήστες για τις δευτερεύουσες εκδόσεις. Ε, βεβαίως είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μειώσει τη γραφειοκρατία εκεί όπου απαιτείται. Ε, και αυτό είναι αναγκαίο, είναι στοιχείο αναγκαίο για τις κεφαλαγορές. Ευχαριστώ τον κύριο Χέ και τώρα δίνω τον λόγο στην ε, κυρία Περβάνς Μπέρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε ούτως ώστε η πρόταση της Επιτροπής να βελτιωθεί σε ορισμένα σημεία και κυρίως ως προς την προστασία των επαγγελματιών επενδυτών των θεσμικών. Θα ήθελα εγώ να είχαμε προχωρήσει περισσότερο και ως προς το, την σύνοψη να το κάνουμε ένα πραγματικό μέσο πρόσβασης για επενδυτές, μη επαγγελματίες, εναρμονίζοντας το περιεχόμενο με αυτό ε, που θα έχουμε στα πλαίσια της νομοθεσίας TRIPS για προϊόντα. Ήταν εκεί μια πρόοδος που θα μπορούσαμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε. Χαίρομαι για την υιοθέτηση ενός ενομερωτικού δελτίου ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτω ώστε να υπάρχει πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις κεφαλαιαγορές που εξαρτώνται από την πολιτική περιορισμένων πιστώσεων τραπεζικών. Ε, χαιρόμεθα για τις συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών και ελεγκτικών αρχών της χώρας καταγωγής και της χώρας διανομής των ενημερωτικών δελτίων. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπέρες. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Στόλογιαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ψηφίσω υπέρ ε, της έκθεσης Γέζεκ και ε, υπέρ ε, οποιοδήποτε μέτρου που στόχο έχει την αύξηση της ε, συμμετοχής της κεφαλαγοράς στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων κατά την έκδοση χρεογράφων ή ομολόγων. Το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να πληρεί τρεις προϋποθέσεις. Θα πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται οι επενδυτές. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τους εκδότες του ενημερωτικού δελτίου και τρίτον, θα πρέπει το ενημερωτικό δελτίο να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα α, αυτούς τους τρεις στόχους και τα τρία αυτά κριτήρια ε, πληρή πρόταση κανονισμού. Ε, προβλέπει με λεπτομέρειες ε, τις πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο, ενώ ταυτόχρονα απλουστεύει την τρέχουσα οδηγία και διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τις επιχειρήσεις που εκδίδουν επιπλέον κινητές αξίες στην αγορά. Και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δέσμευση που ανέλαβε υπέρ της καλύτερης εποπτείας των χρηματαγορών. Επίσης προβλέπει δωρεάν έκδοση πολλών ενημερωτικών δελτίων, ώστε οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση χωρίς επιπλέον κόστος. Σας ευχαριστώ κύριε Στόλογεν. το λόγο ο κύριος Πολ Τάγκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο τελευταίος ε, ομιλητής αυτή την νυχτερινή βάρδια. Θα ήθελα να πω κι εγώ ε, λίγα λόγια. Γιατί πολλές φορές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσκρούν σε διασυνοριακά εμπόδια που εμποδίζουν την πρόσβασή τους στο δανεισμό και η έλλειψη κοινοτικών κανόνων δυσκολεύει την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και χαίρομαι για την ε, αναθεώρηση της οδηγίας και την εναρμόνιση του ενημερωτικού δελτίου. Είναι σημαντικό σημαντικό εργαλείο πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά και είναι σημαντική, σημαντικός ο περιορισμός της γραφειοκρατίας για τις επενδύσεις. Αυτό είναι ένα βήμα προς μια γνήσια ένωση κεφαλαγορών. Φυσικά θα χρειαστούμε ακόμη περισσότερα βήματα και καλύτερη ασφάλεια των επενδυτών. Ίσως κόλλησε αυτό το θέμα στον τριμερή διάλογο εκτός και αν το Συμβούλιο αφουγκραστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μακάρι. Ε, εν πάση περιπτώσει, η ενδιάμεση αναθεώρηση χρειάζεται πιο τολμηρές ενέργειες προκειμένου να έχουμε μια πραγματικά ε, καινούργια γνήσια ε, ένωση κεφαλαιογορών. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω όμως, κύριε Τάγκο, ότι δεν είστε ο τελευταίος ομιλητής στη συζήτηση, γιατί έχουμε και τη διαδικασία Catch και τον κύριο Νότι Μαριά που αυτό θα είναι ο τελευταίο ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την τιμή που μου κάνετε να είμαι ο τελευταίο ομιλητή. Θεωρώ βεβαίω, όπω και όλοι οι συνάδελφοι ότι ο στόχο τη Ένωση των Κέφαλαιων Αγορών είναι να βρεθούν πηγέ χρηματοδότηση κυρίω για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Αυτό σημαίνει διαφάνεια, ενημέρωση του κοινού μέσω του ενημερωτικού δελτίου και οπωσδήποτε η εξάλληψη του γραφειοκρατικού άχθους έχει μεγάλη σημασία ιδίως για δημόσιες προσφορές αξιών κάτω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ. όμως κύριε dombrovskis ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση διότι στο σημείο εννέα της αιτιολογικής έκθεσης αναφέρει ρητά ότι μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδουν τα κράτη μέλη που εκδίδουν οι περιφερειακές οι τοπικές αρχές διεθνείς οργανισμοί που συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη της ένωσης άρα ο esm ο efsf και ενδεχόμενα ο efsm δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν τον παρόντα κανονισμό όπως και η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών. γιατί υπάρχει αυτή η εξαίρεση κύριε dombrovskis; θα θέλαμε μια απάντηση. δεν πρέπει να υπάρξει διαφάνεια και σε σχέση με τις εκδόσεις από πλευράς αυτών των οργανισμών. ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Βάλντις Ντομπρόφσκης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα επ' ευκαιρία να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως τον εισηγητή τον κύριο Γιέζε, καλά και τον προκατοχό του και τους συναδέλφους ε, του που συνεργάστηκαν για την πρόθεση αυτού του θέματος ε, ε, στους τριμερείς διαλόγους και τους ευχαριστώ θερμά για την μεγάλη πρόοδο που σημειώσαμε στις διαπραγματεύσεις. Τώρα προσβλέπω τη συνεργασία και με την ΕΣΠΑ για τα χρονοδιαγράμματα για το ενημερωτικό δελτίο. οπότε θα πρέπει κατεπηγόντως να καταλήξουμε στα εφαρμοστικά μέτρα ώστε να εφαρμοστεί το ενημερωτικό δελτίο από το 2019. Τώρα να απαντήσω στον κύριο Μαριά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα υπόλοιπα θεσμοί που αναφέρατε ανέκαθεν εξαιρούνται σε τέτοιου είδου περιπτώσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Και τώρα θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Πέτρε Γέζεκ, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, δεν μου είχε πει κανείς ότι θα ήταν νυχτερινή απασχόληση η δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαίου αλλά έτσι μας έτυχε σήμερα. Πάντως χαίρομαι που αυτά τα πρώτα στοιχεία της Ένωσης Κεφαλαίου συγκέντρωσαν τόσο ενθουσιώδη υποστήριξη και το, το εκλαμβάνω αυτό σε ένα κοινό επίτευγμα. Και το λέω όχι μόνο από άποψη ουσίας της πρότασης, αλλά επειδή ε, τη σήμερα ημέρα που οι καιροί είναι και μερικοί διστάζουν και κλονίζονται, αυτό το παράδειγμα μας δείχνει περίτρανα ότι οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και τα ε, κοινοτικά θεσμικά όργανα είναι ικανά να συνεργαστούν και να αποφέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ και καληνύχτα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Σίγητα. Ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία της έκθεσης θα λάβει χώρα αύριο. Διακόπτεται η σύνοδος. Θα συνεχιστεί αύριο, Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017, από τις 9 το πρωί. Έχει δημοσιευθεί ε, και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου